Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας με το σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Γαλάζια ανάπτυξη, προαγωγή της αηφόρου ανάπτυξης ε, στις, ε, στα θαλάσσια θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον τουρισμό. Τον προηγούμενο Νοέμβριο πάλι είχαμε τότε αποφάσισαν οι συντονιστές ότι θα γνωρίζουν επ' αυτής της έκθεσης που η πρωτοβουλία είναι της Επιτροπής Τρανς. Η γνωμοδότηση δόθηκε στον κύριο Σαλαβράκο θέμα, που σήμερα θα μας παρουσιάσει ακριβώς το σχέδιο αυτό γνωμοδότησής του. Έχετε αμέσως τον λόγο κύριε Σαλαβράκο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, οι συναδελφοί, οι τομεί τη γαλάζια ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών και του τουρισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστούν ένα πολύ ευρύ πλαίσιο και πολλά θα μπορούσαν να λεχθούν και να γραφούν. Οι τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης είναι πρώτον ο θαλάσσιος και ο παράκτιος τουρισμός, η γαλάζια ενέργεια, η θαλάσσια ορυκτή πόρη, η υδατοκαλλιέργεια και πέμπτον οι γαλάζιες τεχνολογίες. Όπως αντιλαμβάνεστε το έδρος της γνωμοδότησης είναι περιορισμένο και έτσι προσπάθησα να περιορίσω τους τομείς που εμπίπτουν στον τομέα εργασιών της Επιτροπής μας. Η οικονομική κρίση δημιούργησε μια δύσκολη κατάσταση στην Ένωση που αποτελεί μια απειλή αλλά και δυνητικά μια ευκαιρία. Το σχέδιο γνώμη που σας παρουσιάζω τονίζεται ο σημαντικός ρόλος των ωκεανών και της θάλασσας ως τομείς που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά ωφέλη στην ευρωπαϊκή οικονομία παράγοντας ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μέσα από κοινέ συντονισμένες δράσεις μεταξύ άλλων στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας και της ελίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον κλάδο της υδατοκαλλιέργεια που αποτελεί σημαντικό κλάδο της γαλάζιας ανάπτυξης και που συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της παράκτησης κοινότητες. Αναγνωρίζονται τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από την ανάπτυξη σε διάφορους θαλάσσιους τομείς όπως από τις παράκτιες ενεργειακές εγκαταστάσεις ή από την θαλάσσια εξόριξη ορυκτών Τονίζεται ωστόσο η αναγκαιότητα προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντο και των αλλιευτικών πεδίων και η ανάγκη υψίστης προσοχή για την αποφυγή πρόκληση ζημία που μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο και για το συντονισμό των διάφορων δραστηριοτήτων που διενεργούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον κρίνεται πολύ σημαντική η ανάπτυξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού Maritime Spatial Planning και της ολοκλήρωσης διαχείρισης των παρακτήνων ζωνών, απελευθερώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις προοπτικές ανάπτυξης διάφορων θαλάσσιων λεκανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποκλειστικέ οικονομικές ζώνες των κρατών μελών έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη μιας ασφαλούς και αποτελεσματικής γαλάζιας οικονομίας. Μια επιτυχής γαλάζια οικονομία απαιτεί ασφαλή ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνολα για την ανάπτυξη της βιώσιμης αλληλείας, τον έλεγχο, την αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ευβολή του νόμου. Τέλος, τονίζεται η σημασία των παράκτιων περιοχών και του παράκτιου τουρισμού για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ να ακούσω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. gracias, señor Salabracos. Señora Ähm, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνολικά πρέπει να πω ότι είναι μια πολύ καλή γνωμοδότηση αυτή που δόθηκε τώρα από τον κύριο Σαλαβράκο και σας ευχαριστώ για αυτή τη γνωμοδότηση. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την δική μας ομάδα, για την ομάδα Άλντε. Με αυτό το θέμα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ασχολήθηκα. Είναι σημαντικό να βρει κανείς τι είναι καλό σε σχέση με την Επιτροπή Αλληλείας και είναι θετικό για την εκστρατεία, για την μπλε εκστρατεία ακριβώς, για την αηφόρο ανάπτυξη. Κάποια πράγματα είναι σημαντικά που θα ήθελα να συμπληρώσω και θα τα συμπληρώσω και με τροπολογίες και προτάσεις. Πρώτον, βρίσκω πολύ καλό ότι αναφέρετε τις συνέργειες που υπάρχουν. Όταν διάφοροι εμπλεκόμενοι συμπεριλαμβάνονται στην γαλάζια ανάπτυξη. Θα ήθελα εδώ την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική να αναφέρουμε και να εντάξουμε. Δεν είναι πολύ γνωστή, αλλά επ' αυτής βασίζεται η κιανή, η γαλάζια ανάπτυξη. Πρέπει να την αναφέρουμε. Πρέπει να, ε, με την επικοινωνία να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Έχουμε τις ημερίδες θαλασσών, αλλά αυτό είναι λίγο και δεν επαρκεί. Δεύτερο, είναι σημαντικό η πρωτεϊνούχα κάλυψη μέσω ηχθείων, μέσω των ψαριών να προαθεί. Σημαντικό για την κατανάλωση των ψαριών αυτό. Για το σημείο 3 θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι ότι γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο η ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών είναι αναγκαία για την αλληλεία και την έρευνα για τα θέματα θαλασσών να έχουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική έχουμε ένα κονδύλιο στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε και να ανταλλάσσουμε και στοιχεία. Ανταλλάσσοντα στοιχεία υποφελούνται πολύ και στον τομέα αλληλεία βέβαια θα υποφεληθούν. Ένα σημείο 5 ως πρόταση. Θα μπορούσε να συμπληρώσει κανείς λέγοντας ότι στο EMFF υπάρχει για πρώτη φορά ένα κονδύλιο που ε, ξέρω ότι δεν ικανοποιεί όλους αυτό, αλλά είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που καταδεικνύει πώς η πολιτική για την ατυλή αλληλεία είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και της γαλάζιας ανάπτυξης. Σημείο 6. Πολύ καλό το βρίσκω το ότι επισημάνατε τις Διεθνείς Συμφωνίες Αλληλείας. Διαρωτώ με, θα έπρεπε αυτό να ενταχθεί εδώ. Μια όμως ε, και οι συμφωνίες αλληλείας έχουν σχέση και με την πολιτική γειτονία, το βρίσκω σωστό αυτό, το ότι δώσατε συνέχεια με αυτή την πρόταση. Και τελευταίο σημείο, με την, τον παράκτιο τουρισμό, θαλάσσιο τουρισμό, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ και την ε, μικρής κλίμακας βιοτεχνική αλληλεία και αυτό είναι κάτι το οποίο συνδέει αυτά τα θέματα με αυτό το, το ζήτημα. Από την Βόρεια Γερμανία, από την οποία προέρχομαι, οι αλληλείς καβουριών έχουν και μια τουριστική σπουδαιότητα, τουριστική σημασία. Πάνε τουρίστες στις περιοχές τους για να τους δουν και να τους επισκεφθούν. Έτσι μπορούμε λοιπόν και την αηφορία στην αλληλεία με μια τέτοια πρόταση να την προαγάγουμε. Σας ευχαριστώ, μου άρεσε η γνωμοδότησή σας. Σας ευχαριστούμε, κυρία Λεβίν παρακαλώ. Uh, thank you very much, Chair, and uh, thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Σελαβράκο για αυτή την εξαιρετική ε, γνωμοδότηση. Πολλά μπορούμε να πούμε για την ε, μπλε ανάπτυξη. Σίγουρα πάντως δεν είναι απολύτω σαφές τι συμπεριλαμβάνει. Αυτή η έννοια, η έννοια της μπλε ανάπτυξης δεν έχει καθοριστεί επακριβώς. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει πολλά και διάφορα. Γι' αυτό συμφωνώ με την προσέγγιση ε, που ακολουθείτε, να, δηλαδή να συμπεριλαμβάνετε πολλά διαφορετικές πτυχές του ζητήματος στην ομοδότησή σας. Υπάρχουν επίσης όμως και κάποιες ανησυχίες που αφορούν την πλέον ανάπτυξη, την ε, ε, κατάσταση των, του βυθού. Για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι τα δύο τρίτα των υδάτων είναι ε, δεν είναι εθνικά ύδατα και υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ κρατών για τους φυσικούς πόρους, για τους ορυκτούς πόρους, για τους γενετικούς πόρους και για την αλία. Και εκεί υπάρχει μια έλλειψη, δεν υπάρχει ένα ε, πλαίσιο ρυθμιστικό για την ε, εκμετάλλευση αυτών των φυσικών πόρων που βρίσκονται εκτός των εθνικών υδάτων. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε διεθνές επίπεδο αυτό το πρόβλημα, νομίζω, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, της Οργάνωσης ε, Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και οποιοδήποτε άλλο φόρουμ διεθνούς που θα μπορούσε να ε, εντείνει τη διεθνή συνεργασία. Αυτό είναι απαραίτητο διαπιστώνοντας την αυξανόμενη ε, προσπάθεια κρατών να εκμεταλλευτούν αυτούς τους φυσικούς πόρους. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυστηρούς κανόνες για οποιαδήποτε δραστηριότητα εκμετάλλευσης των φυσικών θαλάσσιων πόρων. Ίσως λοιπόν αυτό να μπορούσε να προσθεθεί ως παρατήρηση στην γνωμοδότησή σας. Τώρα στο σημείο 4 που αναφέρεστε στα θαλάσσια σύνορα και την ε, προστασία του περιβάλλοντος, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αυτή, η προσέγγιση είναι μία πιθανή προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση θα μπορούσε να είναι όμως η ενίσχυση της συνεργασίας, δηλαδή να αυξηθεί η συνεργασία στα ζητήματα αυτά. Δηλαδή η συνεργασία μεταξύ κρατών σε περίπτωση περιβαλλοντικής καταστροφής και με τρίτες χώρες, όχι μόνο μεταξύ των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως λοιπόν να είχε νόημα να προσθέσουμε κάποια σχετική διατύπωση. Τώρα στο σημείο 6 που αναφέρεστε στη σύναψη φιλόδοξων διεθνών συμφωνιών για τη βιώσιμη αλληλεία. Ε, συμφωνούμε πλήρως ότι αυτές θα πρέπει να είναι πλήρως εντελώς φιλόδοξες, αλλά όταν τίθεται το ζήτημα του σεβασμού του περιβάλλοντος και της ε, αηφορίας και της βιωσιμότητας, αυτό πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη σε αυτές τις διεθνείς συμφωνίες. Επίση αναφέρεστε στο χωροτεξικό σχεδιασμό, το θαλάσσιο χωροτεξικό σχεδιασμό και την ενιαία πολιτική. Πράγματι χρειάζεται αυτός ο σχεδιασμό να αναπτυχθεί περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που θα διευκολύνει και την κατάρτιση περιβαλλοντικών, ε, αξιολόγησης περιβαλλοντικού αντικτύπου των θαλασσίων δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν προσθετικό αποτέλεσμα, δηλαδή εξόρισξη φυσικών πόρων, η αλληλεία, όλα αυτά ε, έχουν συσσωρευτικό αποτέλεσμα. Ο τουρισμός επίσης, οποιοδήποτε δραστηριότητα έχει επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα πρέπει να έχουμε μια κοινή ε, αξιολόγηση της κατάστασης. Συνολικά πάντως πρέπει να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτή τη γνωμοδότηση και θα ίσως υποβάλω ορισμένε τροπολογίες για να τη βελτιώσω ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. σε ευχαριστούμε κυρία Λεβίν. Η κυρία Γκαρσία Γέρο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλαβράκο για το σχέδιο γνωμοδότησής του εστιάστηκε, επικεντρώθηκε με τέτοιο τρόπο στη γνωμοδότηση που τα πράγματα είναι, πήγαν πολύ σωστά, με το σωστό τρόπο το, τα έκανε. Το να προσπαθήσει κανείς στο μέλλον τώρα να υπάρξει μια νομοθεσία που από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίζει ότι όλες οι οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο περιβάλλον αφενός θα προστατεύουν τους θαλάσσιους πόρους και ταυτόχρονα θα δημιουργούν και μια υφόρο ανάπτυξη μέσω αυτών των δράσεων που θα επικεντρώνεται στις μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές ε, για παράδειγμα. Τα διασυνοριακά προβλήματα που υπάρχουν, το παράνομο εμπόριο ανθρώπων ή ναρκωτικών ή όπλων, όλα αυτά Όλα αυτά μέσω της, των θαλάσσιων μεταφορών να διεξάγονται και πρέπει να αληθούν υπόψη και πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά. Δεν είναι όμως τομέας της αλληλείας. Αυτό θέλω και πάλι να αναφέρω και να, πω, να τονίσω ότι κάνατε μια πολύ καλή έκθεση. Και πέρα από το ότι θα θέσω κάποιες τροπολογίες ως κοιόδης εισηγήτρια της Σοσιαλδημοκρατικής Ομάδας. Πέρα από αυτά θεωρώ ότι οι πιο ουσιώδεις πτυχές συμπεριλαμβάνονται στη γνωμοδότησή σας όπως είναι η οδηγία πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική ή οι οδηγίες για το habitat, τους βιοτόπους. Και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στον ενεργειακό τομέα ότι όλε οι ανθρώπινε δραστηριότητε και οι οικονομικέ δραστηριότητε πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται υπό την πτυχή του να λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι παράγοντες ακριβώς ε, που αναφέρεται. Και να τονίσω στο τέλος ότι είναι αναγκαίο το δυνατόν γοργότερα, πιο σύντομα, να υπάρξει αντίστοιχη νομοθεσία στην οποία θα προβούμε. Είναι πολλές οι δυσκολίες, ε, σπανίζουν οι πόροι, είναι πολύ σπάνια τα κονδύλια, αλλά μέσω από την άλλη πλευρά μιας θαλάσσιας πολιτικής που θα είναι ολοκληρωμένη στο χαρακτήρα της και μέσω ελέγχων από την άλλη πλευρά, ελέγχου των μεταφορών στα θαλάσσια ύδατα, όπου μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο όχι μόνο για την καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας, και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας αλλά και όλες αυτές τις πτυχές που ανησυχούν όλους από, υπό το πρίσμα τουλάχιστον εμένα προσωπικά όπως είναι τα θέματα της ανθρωποεμπορίας, της εμπορίας ανθρώπων ή της παράνομης κυκλοφορίας κεφαλαίων ή και τα θέματα ασφάλειας. στο συγκεκριμένο θέμα της αλληλείας που μας ενδιαφέρει η συνεισφορά αυτής της ε, γνωμοδότησης προς την ε, έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών είναι σημαντική. Θέλω να σας συγχαρώ και πάλι για το έργο που επιτελέσατε με τη γνωμοδότησή σας κύριε Ισηγητά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Βιλάνα παρακαλώ. Θέλω να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Σαλαβράκο γιατί προκαλεί μια συζήτηση θα έλεγα σε ένα σημαντικό θέμα εδώ. Καταρχάς, η κιανή αυτή ανάπτυξη επί της ουσίας θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να δούμε και σε τι κατάσταση είμαστε εμείς για να συζητήσουμε ένα τέτοιο θέμα. Όταν μιλάμε για τη θάλασσα, είναι ένα μέσο από το οποίο περνούν τα εμπορεύματα συνήθω και σπάνια. Ε, eh, Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα εδώ σε σχέση με την αντίληψη που έχουμε για το συγκεκριμένο στοιχείο θα έλεγα. Η προσπάθεια που κάνουμε εμείς τώρα δεν θα έχει αποκλειστικό στόχο βέβαια το θέμα της βιοπικιλότητας, ούτε και τα θέματα τα οποία άπτονται ε, άμεσα ε, και αποκλειστικά με την αλληλεία. Πρέπει όμως να είμαστε κάπως πιο συγκεκριμένοι. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι προσπάθειες τις οποίες έχουμε κάνει και οι οποίες καρποφόρησαν τους τελευταίους μήνες στην Αλληλία να είναι τμήμα της συγκεκριμένης αυτής μορφής ανάπτυξης. Συζητήσαμε σήμερα το πρωί για ένα θέμα όπως είναι η χωροταξία των ακτών και των ίσων κτλ. Πρέπει να δώσουμε κεντρικό χαρακτήρα σε ένα τέτοιο θέμα. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σαν παράδειγμα σε ρυθμίσεις ε, ε, για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η θάλασσα από τα κράτη-μέλη θα έχουμε αποτύχει. Η βάση μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής είναι οι διαφορετικοί κόσμοι που ζουν γύρω από τις θάλασσες να μπορέσουν στα πλαίσια του διαλόγου να οδηγηθούν σε αντίστοιχες οσμώσεις έτσι ώστε να υπάρξει ανάπτυξη, να υπάρξει απασχόληση, να υπάρξει ευφυής χρήση ε, του πληθυσμού των αλλιευμάτων και σε αυτό θα συμφωνήσει μαζί μου και η κυρία Λόδινγκ. Αυτά δεν θα τα πετύχουμε αν δεν υπάρξει σωστό συντονισμό στον τομέα, τον χωροτακτικό θα έλεγα, των περιοχών γύρω από τη θάλασσα. Αλλιώς η προσπάθεια που κάνουμε θα παραμείνει μια θεωρητική, πολιτισμική αν θέλετε προσπάθεια, η οποία δεν θα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. <clears throat> Πιστεύω λοιπόν και θα καταθέσω μια τροπολογία προς την κατεύθυνση αυτή, να υπογραμμίσουμε τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για την χωροτακτική διάταξη αν θέλετε της θάλασσας και των περιοχών γύρω από τη θάλασσα. Έτσι θα ορίσουμε σωστά τις δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στην θάλασσα και οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται με σωστό τρόπο. Γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι ό,τι προσπάθειες και να κάνουμε σε μεμονωμένο επίπεδο, αποκλειστικά στον τομέα της αλληλείας σαν παράδειγμα, ακόμα και με τα νέα επιλεκτικά μέσα, ακόμα και τα νέα δωροφορικά μέσα, αν δεν έχουμε σαν παράδειγμα συγκεκριμένη άποψη για την χρήση της πλατφόρμας την οποία θα έχουμε της θάλασσας δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, νέα ανάπτυξη, ναι και ανάπτυξη, πρώτα όμως οι πολίτες των περιοχών αυτών. Οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι θεματοφύλακες, αν θέλετε, της θαλάσσιας κληρονομιάς, είναι και οι φύλακες, αν θέλετε, αυτής της πολύ σημαντικής πηγής ανθρώπινης διατροφής. Λοιπόν, η γνωμοδότηση αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον, πρέπει να περάσει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις που να αντιμετωπίζουν επιτέλους τα προβλήματα. Έτσι ώστε να καταφέρουμε να υποχρεώσουμε τις μεμονωμένες χώρες να υιοθετήσουν τα μέτρα τα οποία χρειάζονται. Ευχαριστώ κύριε Μιλάνα. Στίβενσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ στον κύριο Σαραβράκου για αυτή την νομοδότηση γαλάζια ανάπτυξη και η βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη νομίζω είναι απαραίτητη. Πάνω το 90% του άνθρακα βρίσκεται στα θαλάσσια υποσυστήματα και τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Μαγκρόβια έλλη. In Europe in particular we have a lot of the latter Uh, Scotland, Εμείς στη Σκοτία έχουμε το 20% αυτών των ε, εκτάσεων των λιβαδικών των θαλάσσιων, των Ποσειδονιών. Ε, θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα τα προστατεύσουμε γιατί οι περιοχές αυτές σορεύουν αν θέλετε και κρατούν ε, δέκα φορές το διοξίδιο του άνθρακα που συγκρατούν τα τροπικά δάση. Αυτό γίνεται στις Ποσειδονίες όπως επίσης και στις περιοχές όπου υπάρχουν υψηλά φύκη. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουμε και τεχνολογικές λύσεις και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να εκμεταλλευτούν ε, τις εκτάσεις αυτές, τις ποσειδονίες αυτές με τρόπους οι οποίοι θα είναι αντίθετοι με το περιβάλλον και κανένας όταν προγραμματίζει τέτοιου είδους μορφές εκμετάλλευσης των θαλασσίων αυτών και παρακτήων περιοχών δεν υπολογίζει τις συνέπειες στο περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να μην καταστρέψουμε τις περιοχές αυτές, τις εκτάσεις αυτές και γι' αυτό λοιπόν η αηφορία είναι το βασικό χαρακτηριστικό της κιανής αυτής μορφής ανάπτυξης. Θα πρέπει εδώ και να προσμετρήσουμε σωστά τις εκπομπές καυσαερίων από τέτοιες δραστηριότητες και ο κύριος Σαλαβράκος είμαι σίγουρος ότι δεν τα αγνοήσει όλα αυτά. Ε, και εγώ ευχαριστώ και πάλι για το θέμα της ολοκληρωμένης ε, θαλάσσιας πολιτικής με απασχολείται και χρόνια. Είμαι και στην Επιτροπή Μεταφορών Πρόκειται επίση και για τη γαλάζια ανάπτυξη και στην Επιτροπή Μεταφορών ω αρμόδια επί τη ουσία κοινοβουλευτική Επιτροπής. Πολύ πρόσφατο είναι ένα κανονισμό για την θαλάσσια χωροταξία και αυτή η πρόταση σχετίζεται πολύ με τα θέματα τη επιτροπή ελληνία. Όλα αυτά θέλω να σα πω ότι τα παρακολουθώ και τα επεξεργάζομαι συνειδητά και στι δύο κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Εγώ εγώ Βόρειο Γερμανίδα θέλω να υπάρξει η αηφορία στην ανάπτυξη. Υπάρχουν διάφοροι τομεί που με τη θάλασσα μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Και λένε όλοι ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους ε, που θα κατοικούν την οικουμένη και πρέπει να δούμε και τον ρόλο των παράκτιων περιοχών και των θαλασσίων δραστηριοτήτων. Πρέπει να διατηρήσουμε την ε, θάλασσα για τις αηφόρες ε, δραστηριότητες για πολλές γενναίες και να μην καταστραφεί. Είναι πολύ σωστό αυτό. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση της ολοκληρωμένης πολιτικής για τις θάλασσες. Εντάξει, είναι ένας τομέας οικονομικός η αλία, όπως και οι παράκτιες ε, τουριστικές δραστηριότητες, οι υδατοκαλλιέργειες, ε, οι θαλάσσιες μεταφορές. Όλα αυτά σε μια ολοκληρωμένη πολιτική για τις θάλασσες πρέπει να διασφαλίσουν την επιβίωση των θαλασσών. Και αυτά είναι σημαντικά για μας στην Επιτροπή Μεταφορών που παρακολουθούμε αυτά τα θέματα, να επικεντρωθούμε με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά και στην Επιτροπή Αλίας επικεντρωνόμαστε με ιδιαίτερο τρόπο σε αυτά τα θέματα, διότι όλα συσχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Θέλουμε να διατηρηθεί αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες σας. Τώρα η Επιτροπή θα λάβει τον λόγο. Κύριε Φρύση έχετε τον λόγο. Thank you. Um, thank you to the ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή για την σωστή αξιολόγηση στην οποία προχώρησε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μας. Ξέρετε ότι είμαστε στο σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη μιας ολόκληρης δέσμης διαφορετικών μορφών δράσης. Στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε το αναπτυξιακό δυναμικό το οποίο ενυπάρχει στην θαλάσσια οικονομία, σε ορισμένες πλευρές της τουλάχιστον, και σχολιάζοντας εδώ να πω ότι σωστά δίδεται μεγάλη σημασία στην πρόταση αυτή και από τους ομιλητές άλλωστε στην αηφορία. Φυσικά και συμφωνούμε με αυτό θα προσπαθήσουμε όχι μόνο να ανοιχνεύσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις θάλασσες, αλλά και να τις διατηρήσουμε για τις επόμενες γενναίες. Αυτός είναι στόχος τον οποίο συμμεριζόμεθα όλοι, ένα στόχος τον οποίο θεωρούμε όλοι πάρα πολύ σημαντικό. Η άποψή σας λοιπόν γύρω από το συγκεκριμένο τομέα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα λάβουμε υπόψη μας τα σχόλια τα οποία κάνατε σήμερα εδώ και την τελική σας έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Σαλαβράκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους οι οποίοι τοποθετήθηκαν πάνω στο σχέδιο της γνωμοδοτησής μου. Βεβαίως ε, ο προσδιορισμός ε, γαλάζια ανάπτυξη είναι εντελώς φιλολογικός η θάλασσα είναι ένας χώρος ζωής εκατομμύρια χρόνια. Όσο υπάρχουν άνθρωποι πάνω σε αυτή τη γη. Και σαν χώρο ζωής, σε ένα χώρο που δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι, έχει παθογένειες, έχει αρρώστιες, έχει βεβαίως και τις καλές στιγμές. Ε, εκείνο το οποίο ε, προσπαθούμε με τη γνωμοδότηση αυτή αλλά κυρίως με την έκθεση επί της ουσίας την οποία κάνει εκ μέρους της ΤΡΑΝ ο συνάδελφος κύριος Δανέλης με τον οποίο είμαι σε άμεση επαφή και στην έκθεσή του περιλαμβάνει τα περισσότερα από όσα συμπληρωματικά εδώ ακουστήκανε είναι να κάνουμε μια συστηματοποίηση για τη βελτίωση των δράσεων μέσα στη θάλασσα. Διότι πλέον ακριβώς για τον λόγο ότι Δημογραφικά η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα μεγάλο πρόβλημα έξαρσης. Δεν ξέρω αν θα είναι το 2059 εκατομμύρια, αλλά σίγουρα το 2080 θα είναι 9 εκατομμύρια, δηλαδή θα αυξηθεί ο πληθυσμός κατά 2,5 περίπου δισεκατομμύρια ανθρώπους, ενώ χρειάστηκε 100 χρόνια για να αυξηθεί κατά ένα. Παράλληλα, λόγω της αυξήσεως του πληθυσμού, αντιλαμβάνεστε ότι η θάλασσα σαν πόρος που προσφέρει ζωή, σαν πόρος που προσφέρει τροφή, σαν πόρος που προσφέρει δραστηριότητα, πρέπει να διασφαλιστεί. Διότι για να ζήσουμε με τα υπάρχοντα μέσα, είτε της γεωργίας, είτε της αλληλίας, είτε των παντός είδους μεταφορών, αλλά και της δημιουργίας ευτυχίας των ανθρώπων με τον τουρισμό, πρέπει να κοιτάξουμε και να βάλουμε ορισμένους κανόνες που να την που να κάνουν την θάλασσα πιο πράσινη. Ε, Αγαπητή κυρία Λέβιν, όλοι είμαστε πράσινοι, έτσι, ε, διότι πλέον ε, είσαστε ένα κίνημα παλιά εσείς. Τώρα είναι μια αναγκαιότητα για όλους μας, δεν ξέρω στο μέγεθος των γνώσεων ή των επιδιώξεων των δικών σας ή αν φτάνουμε, αλλά πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε αντιληφθεί ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στο περιβάλλον σκοτώνουν τους ανθρώπους, θα σκοτώσουν τους ανθρώπους ή τουλάχιστον θα σκοτώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Προσπάθησα λοιπόν να είμαι λακωνικός, να πω όσο το δυνατόν πιο λίγα σε αυτή την έκθεση, εις τρόπον ώστε να μην περιγράφουμε επακριβώς τις δραστηριότητες τις οποίες υποθαλπούμε, αλλά να αφήνουμε περιθώριο να χωράνε μέσα σε αυτές τις δραστηριότητες και άλλες οι οποίες μπορούν να έχουν ένα διάφορο ορισμό στην διαδρομή και την αναγκαιότητα την οποία θα μας δημιουργήσει η εφαρμογή ε, της νομοθετικής πλέον ε, πρωτοβουλίας την οποία θα έχει Κομισιόν. Ε, εγώ θα δεχθώ την οποιαδήποτε τροπολογία διότι ε, έχω πάντα την εντυπώτηση ότι σε αυτή την Επιτροπή μιλάμε πολύ φιλικά και πολύ αποτελεσματικά. Ε, και πιστεύω ότι η έκθεση με τις παρατηρήσεις και τις δικές σας θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Muchas gracias, señor Salabracos. Finalizado el debate, comunicarles que el plazo de presentación de enmiendas a este... Ολοκληρώνοντας την συζήτηση εκπνοή προθεσμίας τροπολογιών είναι 27 Μαρτίου το μεσημέρι 12.00. Περνάμε στο 14 τροποποίηση του ε, κανονισμού σε σχέση με την διατήρηση μέσω τεχνικών μέτρων των ε, πόρων στο Μπέλτ, στη Βατική θάλασσα, στο Σούντ. Υπάρχει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως γνωρίζετε. Ο κύριος Γκρομάτσικ ανέλαβε το θέμα. Σήμερα θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και έχει τον λόγο ο κύριος Γκομπάτσικ, παρακαλώ, πρώτος. Έχει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο κανονισμός τον οποίο συζητάμε στην παρούσα φάση και ο κανονισμός τον οποίο θα συζητήσουμε στη δική μας Επιτροπή συνδέεται με τη λήψη τεχνικών μέτρων που τροποποιεί τον βασικό κανονισμό σε σχέση με την χρήση τεχνικών μέτρων στην περίπτωση αυτών των Belts, των Sound και της Βαλτικής γενικότερα έτσι ώστε να προσαρμοστούν οι κανονισμοί αυτοί στις ρυθμίσεις της Λισαβόνας. Καλύπτει επίσης τις λεγόμενες κατεξουσιοδότηση πράξεις, όπως επίσης και όλες τις άλλες μορφές εξουσιοδότησης οι οποίες δίδονται ή περνούν μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχετικά με το βασικό κανονισμό και με τα τεχνικά μέτρα στα οποία αναφέρθηκα στην προηγούμενη συνάντησή μας, όταν και ξεκίνησε η συζήτηση για τον κανονισμό, δεν μπορώ παρά να αναφερθώ για μια ακόμη φορά επίσης και στο θέμα των απορρίψεων, στο θέμα των εξοπλισμών και της χρήσης των εξοπλισμών των αλλιευτικών. και στα θέματα της λεγόμενης βιομηχανικής αλληλείας και στα θέματα της κατανάλωσης των προϊόντων της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Τα θέματα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν και να προσδιοριστούν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε και οι αλληλείς να μπορέσουν να διατηρήσουν την δουλειά τους και το φυσικό περιβάλλον να προστατευθεί. Αυτή είναι η προσπάθεια λοιπόν η οποία γίνεται. Αν κοιτάξει κανείς ποια είναι η κατάσταση και πώς έχει η κατάσταση στον τομέα της αλίας και αν προσέξει κανείς ακριβώς το πώς λειτουργεί η έκθεση της κυρίας Ρόντους που είναι η βασική μας αναφορά αν θέλετε στο θέμα του μέλλοντος των αλλιευτικών δραστηριοτήτων θα δούμε και θα θεωρήσουμε ότι οι προτάσεις και τις προτάσεις της δικής μου και αυτές οι προτάσεις που κάνω εγώ θα μπορούσαν να θεωρηθούν ε, σαν κάτι το πρόημο, σαν κάτι το πρόωρο. Τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να αφορούν κυρίως το μέλλον της αλλιευτικής πολιτικής, γιατί ακριβώς αυτή η πολιτική θα είναι το κεντρικό σημείο, το κομβικό σημείο, το οποίο θα χαρακτηρίσει τη λήψη των τεχνικών μέτρων ε, και για τα sound και για τα belts και για τη βαλτική γενικότερα. Στην περίπτωση συγκεκριμένα τώρα των απορρίψεων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να πάρει κανείς κάποιες αποφάσεις οι οποίες να λειτουργήσουν δεσμευτικά για το μέλλον και σε επίπεδο επίσης αλλιευτικών εξοπλισμών. Ακόμα και αν το κάνουμε αυτό, θα δούμε ότι τα θέματα αυτά στην ουσία δεν θα συζητηθούν από το Συμβούλιο ή αν συζητηθούν δεν θα γίνουν δεκτές οι προτάσεις αυτές και θα οδηγηθούμε για μια ακόμη φορά σε αδιέξοδο. Γι' αυτό ακριβώς και προτείνουμε αυτά τα οποία προτείνει, συμφωνούμε με αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά αυτό το οποίο λείπει στη συγκεκριμένη περίπτωση από εδώ και πέρα και αυτή τη στιγμή γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας για την αλλιευτική πολιτική είναι οι τεχνικές ρυθμίσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο. Ο κύριος Βαλένσα παρακαλώ. Δεν σας είχα δει πιο πριν. Συγγνώμη. Κύριε Βαλένσα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γκρομπότσικ για την παρουσίαση από πλευρά σας. Όπως και προηγούμενα αναφέρθηκε ότι έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι θέλετε να περιοριστείτε αυστηρά στις διατάξεις συνθήκης Λισαβόνας. Δεν μπορούμε όμως να αμελήσουμε, να ξεχάσουμε ότι πολλά από τα στοιχεία αυτού του κανονισμού θα απαιτηθεί πολύ γοργά μετά τη μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής όταν θα έχει αυτή ολοκληρωθεί να τροποποιηθούν. Είναι πολύ μεγάλες οι φιλοδοξίες λαμβάνοντας υπόψη και τις προθεσμίες για την υποχρέωση όσον αφορά τη Βαλτική για παράδειγμα. Εδώ εννοώ κυρίως την αλλαγή του άρθρου 12 που με τη σημερινή της μορφή ε, καθιστά αναγκαίο το να απορρίπτει κανείς ε, ή όλα τα μικρού μεγέθους ψάρια να να μην τα, να ε, κρατά αλλά να τα απορρίπτει πίσω στη θάλασσα και αυτό θα αναφέρεται και στα ε, ε, δίκτυα τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν καθώς επίσης και στο παράρτημα 4 σε σχέση με τα μάτια των δικτυών, ε, σε σχέση με τις διαστάσεις δηλαδή ματιών δικτυών για να προστατεύονται τα αλλιεύματα. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι έτοιμη με την πρότασή της έγκαιρα, ώστε να υποβληθεί έγκαιρα και να αποφύγουμε προβλήματα με την εισαγωγή απορρίψεων ηχθείων στη Βαλτική. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι οι τριμερείς διάλογοι για την, ε, τον κανονισμό βρίσκονται υπό εξέλιξη. Εξαρτάται από το πότε θα ολοκληρωθεί αυτός ο κανονισμός και τότε θα έχουμε και μετά το σχέδιο αυτού του κανονισμού και το θέμα εμπλοκής στα θέματα αυτά από πλευράς των τριμερών διαλόγων. Εργαζόμαστε λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κατάσταση ως έχει σήμερα Δηλαδή όσον αφορά τη δική μας πρόταση, ποια θα, μορφή θα έπαιρνε και με ποιο τρόπο εργαζόμαστε στην Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων DG Mare με ποιες διατάξεις και ποια άρθρα του κανονισμού που θα αλλάξουν και φυσικά σε σχέση με τη Βαλτική απασχολούμεθα και με αυτό το σκέλος για την άρση όλων των εμποδίων και προσκομμάτων για την εκφόρτωση των ε, αλλιευμάτων και θα πρέπει πολλά πράγματα να αλλάξουν όσον αφορά τις τεχνικές ε, λεπτομέρειες ε, και στοιχεία για όλες τις περιοχές, ακόμα και για τη Βαλτική συμπεριλαμβανομένης, δηλαδή και της Βαλτικής. Αναθεωρούμε λοιπόν μέσα σε αυτή τη διαδικασία όλες τις νομικές πράξεις ε, που ισχύουν και που εφαρμόζονται υπό αυτό το πρίσμα προετοιμάζοντας αυτόν τον κανονισμό. Πώς θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές. Εξάπαντος με μια, πρώτη, με μια συνολική σφαιρική αλλαγή και μεταρρύθμιση καλύπτοντας όλους τους κανονισμούς ταυτόχρονα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να άρουμε όλα τα εμπόδια με μια τέτοια δράση για την εκφόρτωση των αλλιευμάτων π.χ. Και όπως ο κύριος συζητητής, κύριος Κρόμπατσίκα, πιστεύουμε ότι σωστά ανέφερε, ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν πρώιμη η χρονική στιγμή, θα ήταν πολύ πρόωρο να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε μόνο τις τεχνικές διαστάσεις και τα τεχνικά μέτρα μόνο για τη Βαλτική. Εμείς σε σχέση με τις τροποποιήσεις αυτές τις κάναμε για να ευθυγραμμιστούμε μόνο με τις νέες διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Και ακριβώς για αυτό το θέμα θα ήθελα να υποστηρίξω και τον κύριο Γκρόμπατσικ στο αίτημά του από πλευρά της Επιτροπής Αλίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο σημείο, το 15. Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή στα ωφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους, τη χρησιμοποίησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων είναι σε σχέση με τις απόψεις των ε, συναδέλφων με τον εισηγητή που είναι ο κύριος Χάτσον και που πρώτος θα λάβει τον λόγο φυσικά. Έχετε τον λόγο κύριε Χάτσον. Thank you, uh, President. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι. Και πάλι θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να ήμουν παρόν, αλλά ήταν η συνάδελφος και ανέλαβε αυτό που θα έπρεπε εγώ κανονικά να κάνω. Λοιπόν, σήμερα θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο να σας παρουσιάσω το προσχέδιο της έκθεσης και να δώσω την ευκαιρία στα μέλη της Επιτροπής να κάνουν οποιαδήποτε παρατήρηση και να ακούσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρωτόκολλο του Σλαγκόγια που αναφέρεται στην πρόσβαση στους γενετικούς πόρους. Και αναφέρεται συγκεκριμένα στα πλεονεκτήματα που παρέχει η πρόσβαση αυτή γενικά. Εμείς προφανώς προσπαθούμε να εστιάσουμε στον αντίκτυπο που έχει αυτό στην αλία, εάν υπάρχουν τέτοιοι, και να βρούμε τις προφανείς περιοχές ε, που μας αφορούν, για παράδειγμα την αλία, την διαχείριση ε, του αλιεύματος. Ίσως υπάρχουν λοιπόν ε, ανάγκες για έρευνα σε σχέση με την αλία ή με την υδατοκαλλιέργεια στις οποίες να μπορεί να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο αυτό. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην καταγραφή δεδομένων από βιολογικούς πόρους και τη σωστή διαχείρισή τους με βάση της πρόνοιες πρωτοκόλλου. Όποτε αυτές οι, αυτοί οι πόροι έχουν προέλθει από πρωτότυπη έρευνα, αναγνωρίζεται το δικαίωμα των κρατών όταν αυτά τα δεδομένα έχουν προκύψει από, βιολογικούς, ε, από βιολογικές πηγές, από οργανισμούς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό που για μένα δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο Επ' αυτού θα ήθελα να θέσω και κάποια ερωτήματα στην Επιτροπή. Συνεχίζονται και τις, τις, τις ερωτήσεις που είχα θέσει μετά την αρχική παρουσίαση. Γίνεται μια αναφορά ή μάλλον είναι απέτηση τα ε, συμβαλόμενα μέρη στο πρωτόκολλο δηλαδή όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητείτε να έχουν ένα σημείο επαφής, το οποίο θα έχει την αρμοδιότητα της διαχείριση και την ευθύνη της διαχείριση των πόρων αυτών. Τώρα, με βάση την πρόταση της Επιτροπής, προτείνεται να δημιουργηθεί ένα ε, σημείο επαφής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα Αυτό που δεν είναι σαφέ είναι πώς, ποια θα είναι η σχέση αυτού του Ευρωπαϊκού Σημείου Επαφή με τα Εθνικά Σημεία Επαφή. Ποια θα είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων, τι ακριβώ θα κάνει το Σημείο Επαφή τη Κομισιόν σε σχέση με αυτά που θα πρέπει να αναλάβουν τα Σημεία Επαφή στα, ε, στα κράτη-μέλη. Και να αποφύγουμε την αλληλοεπικάλυψη. Τώρα το ζήτημα της γεωγραφικής κάλυψης επίσης ε, τίθεται. γίνεται αναφορά στην εθνική κυριαρχία των κρατών και στο ε, εύρος της ΑΟΣ τους, όχι μόνο για τα 12 μίλια. Άρα τίθεται ένα ζήτημα εδώ. Πέρα από την ΑΟΣ, όταν φτάνουμε στα διεθνή ύδατα, θα μπορούσε κάποιος να θέσει το επιχείρημα ότι ε, η εθνική κυριαρχία θα μπορεί να εκτείνεται και σε εκείνα τα πλοία που είναι νεολογημένα με τη σημαία ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους. Πέρα από αυτές τις παρατηρήσεις, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων για να τις λάβω υπόψη μου. Και με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικά για τα συγκεκριμένα θέματα που έθεσα και αυτές τις απορίες που απομένουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λοιπόν, έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί έχουμε προχωρήσει. Έπρεπε να σκεφτούν ότι μετά από τα τρία πρώτα σημεία θα έρθει και το επόμενο. Τώρα φτάσαμε στο επόμενο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο συνάδελφος ο οποίος θα ήθελε το λόγο. Από πλευρά τη Επιτροπή επίση δεν υπάρχει κανείς. Οπότε κλείνουμε το συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το θέμα χωρίς να τους ακούσουμε βέβαια. Κοιτάξτε, θα μπορούσατε να παρακολουθείτε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται, εν περιπτώσει, η συνεδρίαση. Όπως και να έχουν τα πράγματα, ευχαριστώ τον κύριο Χάτον, σας ευχαριστώ όλους. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη. Αύριο στις 9 έχουμε τους συντονιστές. Ευχαριστώ. Εδώ τα πράγματα